Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μαζί με την Λαμεκέβιν και την Έλενα Βαλατσιάνο θα προεδρεύσουμε αυτήν την ε, συνεδρίαση. Βεβαίως κάθε χρόνο συναντιόμαστε με όλους τους ε, πάνω το βραβείο Σαχάροφ για την ελευθερία και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που σήμερα έχουμε την κυρία Άνισαν Χάινταρ, η οποία είναι η σύζυγος και εκπροσωπεί εδώ τον Ράιφ Μπαντάουι, ο οποίος πήρε το βραβείο Ζαχάροφ το 2015. Δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ ο κύριος Μπαντάουι γιατί όπως και στο παρελθόν βρίσκεται ακόμα στη φυλακή και εκτεί την ποινή του, μια ποινή φυλάκισης για εντελώς ε, αδικαιολόγητους ε, ε, λόγους καταδικάστηκε και βεβαίως αυτό είναι αντίθετο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Σταύρος Λαμπρινίδης, ο ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι επίσης σήμερα μαζί μας και φυσικά η εργασία του είναι εξαιρετικά σημαντική. Εξ ονόματος λοιπόν της ε, Επιτροπής μας τον ευχαριστούμε για την ε, συνεργασία που έχουμε μαζί του αλλά και για τα όσα κάνει εξ ονόματος της Εξωτερικής Υπηρεσίας Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία. Ο κύριος Μπαντάου είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει κάνει πολλά. Εμείς Βεβαίως θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προστασία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Όλα αυτά τα χρόνια το βραβείο Ζαχάροφ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή. Πρόκειται, αν θέλετε, για κάτι το οποίο ξεπερνάει τα κόμματα. Είναι μια συλλογική δέσμευση για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως κάθε φορά με αυτό εκφράζουμε την δέσμευσή μας για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, για όλους όσους πολεμάνε για την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως κάποιοι από εμάς και βλέπω εδώ τον Μικούλαμ έχουν μεγαλώσει χωρίς ελευθερία, έχουν υποστεί αυτούς τους περιορισμούς και γνωρίζουν, μπορούν να μας πούν ακριβώς τι σημαίνει. ποιοι άλλοι δεν έχουν κινδυνεύσει ποτέ. Σε άλλες χώρες βεβαίως κινδυνεύει να επιβληθεί τέτοιος περιορισμός της ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό αγαθό είναι η ελευθερία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ κυρία Χαϊντάρ και θα θέλαμε να εκφράσετε τον θαυμασμό μας και την στήριξή μας στον σύζυγό σας. Υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη στον κόσμο που καθημερινά άνθρωποι πολεμούν για την ε, ανθρωπιά, για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία έκφρασης. Και φυσικά αυτή η μάχη είναι αδιάκοπη. Εμείς ε, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστούν αυτές οι θεμελιώδεις ε, ελευθερίες και ότι βεβαίως χρειάζεται συλλογική δράση και υποστήριξη έτσι ώστε να υπάρχει πρόοδο στον τομέα αυτό της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην υπάρχει καμία υποχώρηση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να σιωπήσουμε όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να μην κάνουμε τίποτα, να παραμένουμε άπλογοι. Ο Μπανκιμών είχε αναφερθεί στην ε, ελευθερία έκφρασης, στην πρόσφυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παρακολούθηση, τα συστήματα παρακολούθησης λέγοντας ότι όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζονται, να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Και βεβαίως στην περίπτωση του Γκραπ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρετε ότι σήμερα η σύζυγος του κ. Μπαντάβη καθημερινά συνεχίζει τις προσπάθειές της και προσπαθεί να συνεχίσει την ε, μάχη της. Είναι πραγματικά μια αξιοθαύμαστη περίπτωση ανθρώπου που πολεμάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μπαλατσιάνα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δύο προσωπικότητες και ομάδες βρίσκονται σε αυτούς τους οποίους υποστηρίζουμε και θέλουμε να δοθεί υποστήριξη είναι η δημοκρατική αντιπολίτευση στην Βενεζουέλα που στηρίζουν τους πολιτικούς κρατούμενους και προσπαθούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση Βενεζουέλα και βεβαίως αυτό πριν τις ε, πρόσφατες εκλογές που βοήθησαν να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα αυτή και ελπίζω αυτό το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών να ληφθεί σοβαρά υπόψη να γίνει αποδεκτό από τον πρόεδρο της χώρας αυτής γιατί πρόκειται για μια δημοκρατική διαδικασία καθώς και τον κύριο Νέμψοφ που όπως ξέρετε εκπροσωπείται από την κόρη του σήμερα εδώ ελπίζω και εκείνος να υποστηριχθεί και την Παρασκευή θα συνεχίσουμε στη Μόσχα με τον Καζιάνοφ ο οποίος είναι ο διάδοχός του στο κόμμα και τώρα έχει το λόγο η Ελένα Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Μπροκ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μπατάουι έκανε ένα έγκλημα. Το έγκλημα ήταν να εκφράσει τη σκέψη του με το λόγο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να επιβληθεί μια τόσο σκληρή ποινή και ανελαίει τα βασανιστήρια. Μας φαίνεται σαν ψέμα, αλλά έτσι έγινε. Δυστυχώς ε, τι έκαναν, τον εξύβρισαν, τον βασάνισαν, τον μαστίγωσαν και η οικογένειά του έφτασε ε, στο σημείο να φύγει από τη χώρα. Και αυτό έγινε μέσω ενός ε, blog. Προσπάθησε να προωθήσει μία δημόσια συζήτηση σε μία χώρα που κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Ο Μπαντάουι ήταν υπέρ της ελεύθερης σκέψης, σκέψης εκεί όπου γεννήθηκε. Φάνηκε όμως αποστάτης. Άνθρωποι σαν το Μπαντάουι, μετριόφρονες άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι μιλούν γαλήνια χωρίς ε, να επιτίθενται, φαίνεται ότι αποτελούν απειλή για αυτά τα καθεστώτα γιατί απλώς είπε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη του άλλου και αυτό δείχνει ότι αξίζουμε. Ζήσε και άσε και τους άλλους να ζήσουν. Σκέψου και άφησε και τους άλλους να σκεφτούν. Και ότι η ελεύθερη σκέψη είναι κάτι το αναπόσπαστο εάν, ε, γιατί διαφορετικά δεν θα προωθηθεί η κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς φυλακίστηκε, γιατί εξέφρασε το φόβο του ότι διανοούμενοι της χώρας του βρέθηκαν ε, εκτός χώρας, μέσα στα πλαίσια της ε, μυσαλλοδοξίας. Και γι' αυτό καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια ε, και χίλιες μαστιγώσεις. Μπορεί να βασανίστηκε, να φυλακίστηκε, προσπάθησαν να τον κάμψουν, να τον εξαφανίσουν, αλλά δεν σκιώπησε, δεν τα κατάφεραν. Και γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ, για να μην ε, καταφέρουν να κάνουν τον Μπαντάουι να σιωπήσει. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας όπως κάναμε και το Φεβρουάριο απονέμοντας ε, το βραβείο Ζαχάροφ το οποίο θα απονεμηθεί επίσημα στην επίσημη πανηγυρική συνεδρίαση της Τετάρτης. Μιλάμε για την άμεση απελευθέρωση ενός πατέρα και ενός συζύγου. Ο Ραΐς αποφάσισε να σταματήσει να τρώει και βρέθηκε στην απομόνωση, σε μία φυλακή απομόνωσης. Η Ενσάφ Χαϊντάρ μετατράπηκε σε ακτιβίστρια, υπερασπίστηκε την ελευθερία και τα δικαιώματα του συζύγου της. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε από εμά θα μπορούσε να κατανοήσει την ε, μεγάλη ε, λύπη της Ενσάφ Χαϊντάρ και το πόσο υπέφερε. Άφησε τα μικρά της παιδιά 11, 10 και 8 ετών. Χρειάστηκε να ε, μεταβεί στον Καναδά που ήταν μια χώρα ξένη για αυτήν. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι πέρασε η ΕΝΣΑΦ, τι μάχες έδωσε. Γνωρίζω ότι όπως της είπε ο Ραΐφ θα επιστρέψει και το πιστεύει η ΕΝΣΑΦ και εμείς το ίδιο. Και βρισκόμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε να τα καταφέρει. Μακάρι το κοινοβούλιο αυτό και όλες οι κυβερνήσεις να βοηθήσουμε την ΕΝΣΑΦ να ξαναβρεθεί με τον ΡΑΙΦ. Αυτοί που είναι ανδροί είναι εκείνοι που παρά το φόβο τους μάχονται και υπερασπίζονται τις ιδέες τους. Υπερασπίζονται εκείνους που είναι μαχητές. Δίνουμε το βραβείο σε έναν ανδρείο και θα το παραδώσει μια πολύ γενναία γυναίκα, η σύζυγός του, η Ενσάφ. thank you, Elena. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Ευχαριστώ, Έλμαρ, για αυτά τα εισαγωγικά ε, που μας ε, είπες ε, είναι εδώ και ο, Σταύρος Λαμπρινίδης εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρία Χαϊντάρα είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας έχουμε σήμερα εδώ αφού αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε τη χώρα σας και να ζητήσετε καταφύγιο στο εξωτερικό είναι πολύ λυπηρό για μας που ο σύζυγός σας τον οποίο υπερασπίζεστε δεν είναι σε θέση να βρίσκεται μαζί μας. Ελπίζουμε ότι θα το καταφέρει στο εγγύς μέλλον. Άοκνα έχετε ε, προσπαθήσει να γνωστοποιήσετε ε, την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει και πρέπει να σας πω ότι έχετε εδώ τους εκπροσώπους των, της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής, ε, ε, Υποεπιτροπής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαντικοί στις χώρες τους που έχουν αγωνιστεί και αυτοί για την ειρήνη και την ελευθερία. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λέει η κυρία Χαϊντάρ, ειλικρινά να σας ευχαριστήσω, ε, γιατί πριν από ένα μήνα όταν άκουσα ότι ο σύζυγός μου είχε επιλεγεί ε, ε, για το βραβείο Ζαγάροφ ε, είχα την αίσθηση ότι ε, άνοιγε μια πόρτα ελευθερίας για τον Ραΐφ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που του δώσατε το βραβείο αυτό. Η επιλογή του Ραΐφ, αυτή η επιλογή που κάνατε μου δίνει πραγματικά μεγάλη ελπίδα ότι θα ακολουθήσει ο δρόμος της ελευθερίας για αυτόν. Σας ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Είμαι πολύ ευτυχής αλλά ταυτόχρονα και πολύ λυπημένη γιατί πραγματικά θα ήθελα να είναι εδώ μαζί μας ο Ραΐφ σήμερα. Θα ήθελα να τον δω να παραλαμβάνει ο ίδιος το βραβείο του. Δυστυχώς όμως ε, δεν είναι εδώ. Ωστόσο τα λόγια σας, αυτά που άκουσα σήμερα, ε, αναπτέρωσαν τις ελπίδες μου. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο Ραΐφ και οπωσδήποτε δεν θα σβήσει ποτέ αυτή η ελπίδα μου. Ευχαριστώ για την τιμή ε, που κάνατε στον Ραΐφ ε, δίνοντάς του το βραβείο αυτό. Πιστεύω ότι το βραβείο αυτό αντιπροσωπεύει πραγματικά το πιο σημαντικό βήμα ε, για την ελευθερία, την απελευθέρωση του Ραΐφ. Δεν είχα ετοιμάσει έναν επίσημο ε, λόγο ε, και θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω για αυτό το πολύ σημαντικό βραβείο. Äh, θα δώσω το λόγο στον ε, Σταύρο Λαμπρινίδη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Dear Insaf, dear Raif. Αγαπητέ Χαϊντάρ, αγαπητέ Ραΐφ, εάν ε, μπορέσετε να μιλήσετε μαζί του, να του μεταφέρετε ε, ότι το βραβείο Ζαχάροφ είναι το πιο σημαντικό ε, βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το σημαντικότερο βραβείο για την ε, ελευθερία έκφρασης στο κόσμο. 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν για το μήνυμα αυτό, για το βραβείο αυτό και επομένως είναι ένα σημαντικό μήνυμα ότι εντός και εκτός της Ευρώπης κάθε χρόνο δεσμευόμαστε εμείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ελευθεροτυπία, για την ανεξιθρησκεία, ε, για την επάυση των βασανιστήριων και των σωματικών ποινών αλλά και κάθε μορφής κατάχρησης. Ελευθερία του συνεταιρίζεστε και πάνω απ' όλα αυτό το βραβείο είναι ένα μήνυμα ότι ε, κάθε ένας από μας εδώ στην Ευρώπη είμαστε δεσμευμένοι ε, να προστατέψουμε κάθε έναν ξεχωριστά που υπερασπίζεται και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου της γης. Το γραφείο Ζαχάροφ ε, εστιάζει την προστοχή της ε, Ευρώπης στην συγκεκριμένη περίπτωση στον Ραΐφ τον, ε, στις 9 Ιανουαρίου ε, η Φεντερίκα Μογκερίνη, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, είχε ήδη ε, υπενθυμίσει σε δήλωσή της την βασική και σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον οποιασδήποτε κατάχρησης και αναφερόμενη συγκεκριμένα στον ΡΑΙΦ σε δεύτερη ανακοίνωσή της ε, στις 8 Ιουνίου όταν επιβεβαιώθηκε ε, από, την, ε, το δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας η ποινή του Ραΐφ σε δεύτερη λέω δήλωσή της υπογράμμισε την σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του φυλακισμένου σε περίπτωση που φυλακιστεί. Ε, ο σύζυγός σας μαστιγώθηκε τον μήνα Ιανουάριο ε, και αυτό προκάλεσε ε, μεγάλη απογοήτευση σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν υπάρξει θετική εξέλιξη Ε, αυτή είναι ότι ε, για λόγους υγείας ε, δεν εφαρμόστηκε, δεν εκτελέστηκε το υπόλοιπο της ποινής. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι ε, να ε, σταματήσει ε, τελειωτικά ή να αναιρεθεί μάλλον και ανασταλεί τελειωτικά η εφαρμογή της ποινής και βεβαίως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρξει άφεση και σταλεί τελειωτικα η εφαρμογη της ποινης και βεβαιως θα συνεχισουμε την προσπαθεια απο πλευρα της ευρωπαικης ενωσης ετσι ωστε να υπαρξει αφεση και χαρη Γνωρίζουμε ότι η Σαουδική Αραβία παίζει σημαντικό ρόλο πολιτικό και θρησκευτικό ε, ε, στον ε, μουσουλμανικό κόσμο. Παρακολουθούμε όλοι ε, τις ε, ε, εξελίξεις σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένα άτομα στο βασίλειο αυτό. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι ακτιβιστές οι οποίοι μάλιστα όταν συνελήφθησαν ήταν ανήλικοι έχουν ε, τύχη της μεγάλης μας προσοχής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες. Ωστόσο, πέρα από τα, τους μεγάλους ε, τίτλους ε, με τους οποίους αναφέρθηκε το δικαίωμα των γυναικών να οδηγούν υπάρχουν ακόμα ε, πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων κυρίως όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, όσον αφορά την ανεξιθρησκεία, όσον αφορά την, το δικαίωμα του συγκεντρώνεστε και του συνεταιρίζεστε και βεβαίως όσον αφορά την θανατική ποινή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι χρειάζεται περισσότερος και όχι λιγότερος διάλογος με τις χώρες του κόλπου και τη Σαουδική Αραβία. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι η Σαουδική, Αραβία, η Σαουδική Αραβία θα οικειοποιηθεί όλη αυτή τη διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, βεβαίως το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι γυναίκες ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές φυσικά και δεν το αγνοώ και δεν το παραβλέπω είναι κάτι πολύ ε, θετικό. Ωστόσο, μία γυναίκα ε, ε, από τη Σαουδική Αραβία δεν μπόρεσε να ψηφίσει γιατί αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο ε, στον Καναδά. Γιατί λόγω του ότι ο σύζυγός της εξέφρασε ελεύθερα την θέση του και την άποψή του, εκείνη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της και εκείνος, ο σύζυγός της, δεν μπορούσε να ψηφίσει ευελπιστώ ότι αυτή η οικογένεια θα επανενωθεί σύντομα για το καλό τους, για τον καλό των παιδιών τους, αλλά και ε, στο όνομα της αξιοπρέπειας και της ε, ε, ανθρωπιάς. Εν σάφ, και εμείς θα επιθυμούσαμε να είναι σήμερα ο Ραΐφ εδώ. Ωστόσο είσαι εσύ σήμερα εδώ στη θέση του. Δεν ζήτησες να είσαι θαραλέα, δεν ζήτησες να αφιερώσεις τόσα χρόνια της ζωής σου για να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο ε, ε, για την περίπτωση του συζύγου σου επιδιώκοντας την ε, απελευθέρωσή του τα παιδιά σου δεν ζήτησαν να περάσουν αυτά που περνούν ωστόσο στάθηκες όρθια με θάρρος και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που σε έχουμε σήμερα μαζί μας και ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και σίγουρα θα συμβάλλει, θα βοηθήσει το βραφείο Ζαχάροφ έτσι ώστε να δοθεί δημοσιότητα στην ε, περίπτωση του συζύγου σου έτσι ώστε η ευτυχία να ξαναέρθει στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for, um, Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Αλίο Μαρή που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, με την Αραβική Χερσόνικο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο μπορώ με αυτόν τον τρόπο να ευχηθώ καλώς στο Κοινοβούλιο στην υψηλή προσκεκλημένη μας. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε προσκεκλημένες γυναίκες από τις χώρες του κόλπου, από την Σαουδική Αραβία που εκφράζουν τις απόψεις τους και παρουσιάζουν την ζωή στις χώρες τους. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πραγματικός διάλογος γιατί νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο εξελίσσονται και προοδεύουν οι καταστάσεις. Έχουμε οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία και πολλές φορές αυτές ακολουθούνται με άγνοια της πραγματικότητας όσον αφορά τι συνήθειε και τον πολιτισμό και τον μεν και τον δε. Και νομίζω ότι με το διάλογο μπορούμε να έχουμε καλύτερη κατανόηση και ενδεχομένως πρόοδο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όπως και η Ευρώπη πρέπει να εκφράσει τις αξίες της, να ακούσουμε τις αξίες των άλλων. Σας εύχομαι λοιπόν καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά Ελπίζω να σταματήσουν οι δοκιμασίες που εσείς και τα παιδιά σας γνωρίσατε τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε και μπορείτε να μεταφέρετε τις επιθυμίες που εκφράζει η Ευρώπη στον, στο περιβάλλον σας. Ελπίζουμε ο σύζυγός σας να απελευθερωθεί σύντομα. Thank Τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες, ε, ένα ομιλητής αναομάδα και θα κάνουμε το γύρο. Πρέντα, ο κύριος Πρέντα για το ΕΛΚ. Παντσέρι στη συνέχεια για τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ να ευχαριστήσω τον κύριο Ενσάφ Χαϊντάρ που είναι εδώ ε, σήμερα μαζί μας και όλη την εβδομάδα για να μιλήσουμε για την περίπτωση του Ραΐφ Μπαντάουι και να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ που δεν μπορεί να ε, παραλάβει ο άνδρας της. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Λαμπρινίδη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποδίδεται το βραβείο Σαχάροφ, Σαχάροφ στον ε, κύριο Βαντάουι γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο και η τήρησή τους. Κανένας δεν πρέπει να ε, φυλακίζεται ή να υφίσταται βασανιστήρια επειδή εξέφρασε τη γνώμη του. Το βραβείο Σαχάροφ... Ε, έχει μια συμβολική αξία της ελευθερίας και του θάρρους ανά τον κόσμο. Πέρα από τη συμβολική σημασία θα θέλαμε να υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις για την ενδεχόμενη απελευθέρωση του ε, Μπατάουι. Ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ το είχε εκφράσει αυτό νωρίτερα όταν η κυρία Μπατάουι στις 6 Μαΐου τον συνάντησε. Τέλος θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Λαμπρινίδη και με τη συνάδελφό μου, την κυρία Αλιό Μαρή, για την ανάγκη συζήτησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σαουδικής Αραβίας και αυτό το είδαμε μέσα στα πλαίσια της συνάντησης εκπροσώπων της Σαουδικής Αραβίας στην ΑΦΕΤ. Ελπίζω να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατόν ο Ραϊφ Μπανταουή. Ο κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ. Το άρθρο 19 της ε, Παγκόσμιας ε, Δήλωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται στην ε, ελευθερία έκφρασης όλων των ανθρώπων μιλάει για τη δύναμη του λόγου που δεν γνωρίζει σύνορα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό το άρθρο, γιατί ε, για μας είναι ο φάρος που θα πρέπει να μας καθοδηγεί εκεί ακριβώς όπου παραβιάζονται και ακυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από αίτημα της ε, ε, ομάδας μας απέδωσε το βραβείο στον ε, Ραϊφ Μπανταουή, το οποίο θα παραλάβει η σύζυγός του. Ε, πρόκειται για έναν φυλακισμένο λόγο πολιτικών πεπιθήσεων, γιατί ετάχθη υπέρ της ελεύθερης έκφρασης. Και γι' αυτό ακριβώς στις 12 Φεβρουαρίου το Κοινοβούλιο συνέταξε ένα ψήφισμα υπέρ του Μπαντάουι όπου αμφισβητήσαμε τη στάση της Σαουδικής Αραβίας και είπαμε ότι θα πρέπει να τον απελευθερώσει. Η χώρα αυτή έδωσε τη δυνατότητα ψήφου στις γυναίκες, στις περιφερειακές εκλογές, αλλά είναι πολύ μακριά από τις ε, παγκόσμιες προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε τις συμφωνίες μας με το Ριάντ, γιατί δεν είναι ένα αξιόπιστο καθεστώς ως προς τις δεσμεύσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μας πρόκειται για ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη υποχρέωση απελευθέρωσης του Ραϊφ Μπαντάουι και την εξασφάλιση για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Thank, thank you very... Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Charles Τάνοκ από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ενσάφ Χάινταρ, σας καλωσορίζω θερμά από την ομάδα μου το ECR που είχε, που είχε θεωρήσει εξ αρχής θα πρέπει να απονεμηθεί το βραβείο στον σύζυγό σας. Θεωρούμε ότι η φυλάκιση είναι κάτι το ανέντιμο και το μη αναλογικό και ζητήσαμε την ε, απελευθέρωσή του. Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας μας ε, προκαλεί, προκαλεί τη Δύση και τις δυνάμεις της δύση. Εμείς θεωρούμε ότι ε, εφαρμόζει το νόμο της Σαρία με θανατικές ποινές και κατά των ανηλίκων όπως συνέβη με έναν ανήλικο Σιήτη στη ε, Σαουδική Αραβία. Ε, επίσης, ο σαλαφισμός της Σαουδικής Αραβίας ε, δείχνει ότι είναι άτεγκτος διότι κανένας δεν μπορεί να ανοίξει καν εκεί και να λειτουργήσει χριστιανική εκκλησία. Άρα έχουμε να κάνουμε και με μία διάσταση της ε, εξωτερικής πολιτικής και πιστεύω ότι ο άνδρας σας, η υπόθεση Μπαντάουι κινείται πέρα των συνόρων του Περσικού κόλπου και αφορά και τα Δυτικά Βαλκάνια και το κέρας της Αφρικής. Γι' αυτό χαιρετίζουμε το θάρρος του κυρίου Μπαντάουι και νομίζω ότι η κυβέρνηση του Ριάντ δεν θα πρέπει απλώς να ε, παραχωρήσει την ψήφο στις γυναίκες για περιφερειακές εκλογές. Ίσως θα πρέπει να κινηθεί προς τον 21ο αιώνα, δηλαδή να επιτρέψει στις γυναίκες να οδηγούν. Επίσης, από όσο γνωρίζω, στην Ιεμένη γίνονται ε, ανεξέλεγκτοι βομβαρδισμοί από την Σαουδική Αραβία κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ιδιαίτερα να μην βομβαρδίζονται περιοχές όπου διαμένουν χούτι. Ελπίζω να ανοίξουν τα μάτια πολλών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας γιατί έχουμε εμπορικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το business as usual. Θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να δεχτεί σοβαρές μεταρρυθμίσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ ε, κύριε Χάινταρ που σας ε, ε, βλέπω, κυρίως που θα συμφωνήσω με τον κύριο Λαμπρινίδη όταν είπε ότι μας εμπνέεται γιατί αποτελείται την αιχμή του δόρατος των γυναικών στη Σαουδική Αραβία. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για να γνωστοποιήσει το θέμα του συζύγου σας Ραϊφ Μπατάουι ε, ε, ελπίζουμε πραγματικά ότι και αυτός ε, και εσείς θα μπορέσετε να ξαναβρεθείτε για το καλό των παιδιών σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Χαιρόμαστε γιατί στην Σαουδική Αραβία είναι η κατάσταση ιδιαίτερη και μερικές φορές ξεχνάμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι γιατί μαζικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ομόφωνα ψήφισε υπέρ της υποψηφιότητας ε, του ε, συζύγου σας. Αυτό που θέλουμε είναι και στο Ιράν και στην Σαουδική Αραβία, στη Βενεζουέλα, στη Συρία, οπουδήποτε ε, να έχουν τη δυνατότητα όλοι να ψηφίζουν, να έχουν τη δυνατότητα όλοι να μιλούν ελεύθερα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε, λαμβάνοντας υπόψη υπήρχαν κάποιες πολιτιστικές διαφορές ε, να μην έχουν όλοι τα ίδια ε, δικαιώματα. Ε, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε κατάσταση όμως βλέπουμε ότι ο σύζυγός σας δεν εκάμφει ούτε από τη, τα βασανιστήρια, ούτε από την φυλάκιση, ούτε από τις σκληρές ποινές μετά από τις 50 ε, πρώτες ε, βουρδουλιές, από τις χίλιες που θα έπρεπε σύμφωνα με την ε, ποινή ε, να ε, ε, λάβει. Σταμάτησε η εκτέλεση της ποινής, η οποία όμως, την οποία η Σαουδική Αραβία ήθελε να συνεχίσει και θα ήταν συνώνυμη της θανατικής ποινής. Κατά την άποψή μου, φιλελευθερισμός σημαίνει να μπορεί κανείς να ζει με ελευθερία και επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά την στην ε, Σαουδική ε, Αραβία. Ε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε μία, ένα τμήμα του, της θρησκείας να θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια και επομένως να πολεμάει την άλλη, το άλλο τμήμα. Ε, δεν είναι ε, δυνατόν να αφήσουμε ε, να μην υπάρχει ισοδικία για όλους και επίσης ξέρουμε ότι τους τελευταίους ε, μήνες ε, η κατάσταση στην ε, Σαουδική Αραβία ελέγχεται όλο και περισσότερο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η εξαγωγή της ριζοσπαστικής και ακρεφνούς πολιτικής και ιδεολογίας, η υπόθαλψη του διχατισμού πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο και εμείς είμαστε στο πλευρό όλων των bloggers, όλων όσων μιλούν ελεύθερα, των άθεων, των γυναικών. Είμαστε στο πλευρό όλων αυτών. Δεν είναι δυνατόν οι ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ένα αμάλγαμα ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν ε, και τους τζιχαντιστές που τρομοκρατούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά από την ομάδα Γκουε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή για μας κυρία Ιντάρ που σας έχουμε σήμερα μαζί σας. Βεβαίως και προφανώς ε, θα προτιμούσαμε να έχουμε μαζί μας το σύζυγό σας. Τον σύζυγό σας που καταδικάστηκε γιατί είχε εγκληματίσει λέγοντας ε, την αλήθεια ή εκφράζοντας ελεύθερα τις σκέψεις του. Ε, ε, από το 2012 είναι φυλακισμένος και σήμερα ξεκίνησε και απεργία πείνας. Στέκεστε στο πλευρό του. Είσαστε κι εσείς θαραλέα όσο και εκείνος. Και μέσα από αυτόν χαιρετίζουμε ε, όλους όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί γιατί έχουν εκφράσει τις ιδέες τις ε, ιδέες τους. Ο Ασάν Φαγιάντ το Νοέμβριο ε, καταδικάστηκε ε, σε, στη θανατική ποινή. Ε, είναι ποιητής ε, Παλαιστίνιος και μέχρι πριν λίγο καιρό εκπροσωπούσε την Σαουδική Αραβία. Ε, στην ε, ε, ποιητική Biennale. Επίσης έχουμε και άλλη περίπτωση ανθρώπου ο οποίος καταδικάστηκε στην θερατική ποινή μέσω σταυρώσεως γιατί τόλμησε να εκφράσει την άποψή του. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε πλέον την κατάσταση αυτή σε μια χώρα με την οποία εμπορεύονται οι χώρες μας. Ε, πρόκειται ε, η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα η οποία ε, έχει κάνει, πολλά είναι υπεύθυνη για τον βομβαρδισμό των γεμενητών είναι υπεύθυνη για, την, για τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ελευθερία και οι οποίες πρώτη φορά πήγαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο, έφτασαν στις κάλπες και 900 γυναίκες είχαν το θάρρος να είναι υποψήφιες αυτές τις ε, εκλογές. Μία γυναίκα εξελέγει, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να χαιρετήσουμε τουλάχιστον αυτό το ε, βήμα το οποίο έγινε. Αγαπητή κυρία, είναι σύμβολο ο σύζυγός σας, σύμβολο όλων των καταπιεσμένων ε, στη Σαουδική Αραβία αλλά και στις ε, γειτονικέ χώρες ε, σε αυτή την περιοχή του κόσμου που είναι από τις χειρότερες όσον αφορά τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Ευελπιστούμε ότι οι χώρες αυτές θα αλλάξουν και δεν θα είναι πλέον, δεν θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτές τις βάρβαρες μεθόδους. Όπως και ο κύριος Τάνοκ πιστεύω και εγώ ότι οι εμπορικές σχέσεις με την χώρα αυτή δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν και το λέω εγώ που είμαι Γαλλίδα. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να χαιρετήσω το θάρρος σας και να σας εκφράσω την ε, ικανοποίησή μας ε, γιατί είστε σήμερα εδώ. Thank you very much. And we have the Barbara Lochbieler for the Greens, followed by... Η Μπάρβαρα για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χάινταρ που ήρθατε σήμερα εδώ. Η πράσινη ομάδα πραγματικά θέλει να σας εκφράσει την εκτίμηση προσωπικά σε εσάς αλλά και σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί σας για να μπορέσετε να απελευθερώσετε το σύζυγό σας. Νομίζω ότι με πολύ έξυπνο τρόπο και πολύ θάρρος έχετε ξεκινήσει αυτήν την μάχη. Βεβαίως ξεκίνησε σήμερα όπως ε, μάθαμε η απεργία πείνας του Ραϊφ Μπανταουή και η δική μας υποστήριξη δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει αλλά σίγουρα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή όλων στην κατάσταση στη δική Αραφία. Υπάρχουν όπως ξέρετε καταδίκες, εκτελέσεις, κακομεταχείριση, βασανισμοί και βεβαίως ε, πάρα πολύ σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον ποινικό κώδικα της ε, χώρας σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μία λίγο διαφορετική πολιτική έκφραση μπορεί να καταδικαστεί, να τιμωρηθεί με βασανιστήρια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι ακτιβιστές και υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακιστεί και έχουν καταδικαστεί σε 10-15 χρόνια επειδή παραδείγματο χάρη δεν δείχνουν σεβασμό ή αρκετό σεβασμό προς τις ε, αρχές του κράτους. Είναι λοιπόν σαφείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα να κάνω μια έκκληση εδώ στην κυβέρνηση αυτής της χώρας ότι πραγματικά ο Ραΐφ Μπαντάουι θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση καθώς και όλοι οι άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι που σαπίζουν στις φυλακές. Thank you. The next speaker will be... Ευχαριστώ. Ο Ιγνάσιο Κοράου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την φιλοξενούμενή μας ευχαριστώντας την ε, για αυτόν τον αγώνα που δίνει για τα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω ότι μέσα από αυτό το βραβείο Ζαχάροφ και την αναγνώριση ε, που ε, δίνεται στον ε, κύριο Μπαντάουι. Ελπίζω ότι ε, θα ε, απελευθερωθεί. Δεν το πολυπιστεύω, αλλά ελπίζω. Ε, στις σχέσεις μας με, την Ευρωπαϊ... με τη Σαουδική Αραβία πραγματικά εκφράζεται όλη αυτή η παράνοια των εμπορικών σχέσεων με την... Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει σχέσεις με μια χώρα που είναι από τους χειρότερους παραβιαστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που έχει ένα από τα χειρότερα ρεκόρ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δυστυχώς έχουμε και ένα ε, χάρτη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά μένει κενό γράμμα. Ε, η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Ραΐφ Μπαντάουι είναι, αντιπροσωπεύει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή με χιλιάδες ε, πολιτικούς κρατούμενους, ε, με γυναίκες που καταπιέζονται, με ανθρώπους που δεν μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Ε, αυτή η Σαουδική Αραβία που δεν μπορεί να την αγγίξει κανένας γιατί μαζί με τους άλλους μονάρχες των κρατών του κόλπου έχουν παρεδώσει οικονομικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε σήμερα το βραβείο Ζαχάροφ στον Μπαντάουι αλλά σήμερα ακριβώς έφυγαν βόμβες ε, και ε, για την, από την Ιταλία για να χτυπήσουν ε, τους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους. Ο συνάδελφος Φαντζέρη ωραία τα είπε προηγουμένως, ωστόσο εκπροσωπεί την, τον κυβερνών κόμμα στην Ευρωπαϊκή, στην Ιταλία. Και ε, ο, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός του ε, βγάζει ωραιότατες φωτογραφίες selfies ε, με τους μονάρχες της Σαουδικής Αραβίας η διεθνής κοινότητα ασύνεκτα προχωράει όσον αφορά ε, τις σχέσεις της με την ε, Σαουδική Αραβία. Ο Ραΐφ Μπαντάουι ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπροστά από το μεγάλο τζαμί ε, μαστιγώθηκε 100 φορές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε απλώς και να λέμε ό,τι γίνεται. Θα πρέπει να συμμετέχουμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να μιλήσουμε ε, για αυτούς που συστηματικά ε, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Tokesh from the EPP Group. Ο Τόκες από το ΕΛΚ. Dear Chairman, Chairwoman. Αγαπητοί συμπρόεδρη, κυρία Ένσαφ Χαϊντάρ, Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ε, συμπάθειά μου προς την κυρία ε, Ένσαρ και την ε, αλληλεγγύη μου για την κατάσταση, για την οικογενειακή σας κατάσταση. Από το 88 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία σκέψης εκείνων που συνεισέφεραν ε, μαχόμενοι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ραϊφ Μπαντάουι προώθησε ε, αυτή τη σκέψη στη Σαουδική Αραβία, προσπάθησε να διαφωτίσει την κοινωνία του και να κατατροπώσει την άγνοια. Αυτό του στήχησε την ελευθερία του. Προώθησε και υπερασπίστηκε τις μειονότητες και τις γυναίκες καθώς και τους ελεύθερα σκεπτόμενους. Γι' αυτό ακριβώς το απενεμήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ. Μέσω του βραβείου ζητάμε από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας άμεσα και χωρίς όρους να τον απελευθερώσουν και να σταματήσουν την περαιτέρω μαστίγωσή του. Επίσης ζητάμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων γιατί άσκησαν το δικαίωμά τους για ε, την ελεύθερη σκέψη, υπέρ της ελεύθερης σκέψης στη χώρα τους. Το Σαββατοκύριακο είδαμε να διαγράφεται μια ιστορική ε, δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία. Οι γυναίκες για πρώτη φορά, περιορισμένα βέβαια, πόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγην στις δημοτικές εκλογές. Βέβαια, οι γυναίκες ε, δεν έχουν ε, πλήρη δικαιώματα. Ελπίζουμε όμως αυτό να αποτελέσει αντικείμενο μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν πραγματικά δικαιώματα. Επειδή η Αραβική Άνοιξη οδήγησε σε απογοήτευση Ας ελπίσουμε ότι ο Ραΐφ Μπαντάουι και οι πρόσφατες εκλογές να προωθήσουν πραγματικά τον κοινωνικό διάλογο και την, τον διαφωτισμό στη, στον αραβικό κόσμο. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της ε, τρέχουσας διαδικασίας και ελπίζουμε να μπορέσει να απελευθερωθεί και να εκφράσει ελεύθερα τη σκέψη του. Um, Richard Howitt for the S&D Group. Richard Howitt, S&D, ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΝΣΑΦ. Ε, ήρθαμε σε επαφή μαζί σας τον Καναδά και σας φιλοξενήσαμε στις Βρυξέλλες. Ε, μας τιμά το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ αυτή τη βδομάδα και σε κάθε ευκαιρία ε, σας υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε μεγάλη μάχη για το ΡΑΙΦ, για την ελευθερία την προσωπική του και την ελευθερία έκφρασης της χώρας σας. Η ε, απόδοση του βραβείου Ζαχάροφ δείχνει ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ότου απελευθερωθεί ο Ραΐφ. Θεωρήθηκε ότι προσέβαλε το Ισλάμ. Όχι όμως, δεν το έκανα αυτό. Είναι υπέρ της ελεύθερης σκέψης. Θεωρούμε ότι είναι όνειδος το ότι ε, σπηλώθηκε ο ίδιος γιατί τήρησε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε η αυτού μεγαλειώτης πραγματικά να ε, αποδώσει χάρη στον άνδρα σας. Εν σαφ. Λάβατε το βραβείο Swiss Free Thinker. Σήμερα ε, λαμβάνετε το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά αυτό που θέλετε πραγματικά είναι η ελευθερία του συζύγου σας. Θέλετε να ε, αντιμετωπίσετε αυτή την βαρβαρική φυλάκηση. Χαιρόμαστε γιατί επικοινωνήσατε μαζί του και σας είπε ότι χαίρετε που έλαβε αυτό το βραβείο. Ελπίζουμε να ελαφρύνουμε τον πόνο του και τον δικό σας πόνο και τον πόνο των παιδιών σας επειδή αποχωριστήκατε τον άντρα σας. Ενσάφ γράψατε ένα βιβλίο «Ελευθερία για τον Ραΐφ Μπαντάουι, την αγάπη της ζωής μου». Αυτή τη βδομάδα ε, τιμούμε την αγάπη σας προς Αυτόν, τον τιμούμε και τον ίδιο, απονέμοντάς του αυτό το βραβείο. Ε, τιμούμε τη ζωή την ίδια. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Θάσου Βίσος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ένσα Φαϊντάρ, κύριε Λαμπρινίδη, κυρίε και κύριοι. Είναι μια πολύ συμβολική ημέρα σήμερα. Στις 14 ε, Σεπτεμβρίου πριν από πάνω από 20 χρόνια πέθανε ο Αντρέη Σαχάροφ μετά από την σύλληψή του, την ε, εξορία επί χρόνια. Πέθανε στο σπίτι του και η ομιλία την οποία έπρεπε να προσφωνήσει στο Ρωσικό Κοινοβούλιο τελικά δεν εκφράστηκε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο περιορισμός της ελευθερίας είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα και βλέπουμε εδώ στην Ευρώπη ότι ο θάνατος του Μπόρις Νέμψχο, ο οποίος προσπάθησε πραγματικά να σταματήσει την επίθεση από του Κρεμλίνου και πολλές ζωές χάθηκαν στη Συρία, στο Ιράκ και αλλού το 2015 σε άλλες αραβικές χώρες. Βεβαίως αυτοί δολοφονήθηκαν από διχαντιστές, από δικτάτορες. Όλοι αυτοί οι οποίοι πνίγηκαν στη Μεσόγειο γιατί προσπαθούσαν να διαφύγουν από την τραγική τους μοίρα. Απ' την άλλη το 2015 ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες με την νίκη της αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα. Όσον αφορά λοιπόν τη Βενεζουέλα βλέπουμε ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα Αντίθετα, βλέπουμε την Σαουδική Αραβία, στην οποία η κατάσταση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Δύσκολες ημέρες και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Για μένα αυτά τα θετικά μηνύματα δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν νόημα και αυτοί πραγματικά που συνεχίζουν να πολεμούν αξίζει να τους δίνεται η ελευθερία. Θα ήθελα λοιπόν εξ ονόματος ε, της ομάδας των φιλελευθέρων να στηρίξω τον Ράιφ Πατάουι καθώς ε, και όλες τους τις προσπάθειες τις οποίες βεβαίως θέλουμε να συνεχίσουμε να ενταρρύνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ ονόματος, ή Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ ονόματος των Πρασίνων. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω ε, και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Συναντηθήκαμε ορισμένους ε, μήνες πριν με εσάς και το Ραΐφ όταν έλαβε βραβείο ο Ραΐφ από το Δήμο του Στρασβούργου. Δεν ξέραμε τότε αν ήταν υποψήφιος, τότε η απόφαση ελήφθη μετά και χαίρομαι που ήρθατε εδώ. Τότε είχαμε ελπίσει ότι θα μπορούσε να παρευρίσκεται και ο Ραΐφ μαζί σας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δυστυχώς, αλλά ελπίζω επειδή ακριβώς είσαστε, θα είσαστε εσείς εδώ και με βάση του διεθνούς τύπου θα πιέσουμε την κυβέρνηση να του αποδώσει χάρη και στον Μπουλακαΐρ που έχει προαναφερθεί και τόσων άλλων που είναι φυλακισμένοι στις φυλακές της Σαουδικής Αραβίας διότι τόλμησαν να επικρίνουν το καθεστώς γιατί τόλμησαν όπως ο Μοχάμετ Αλνίμερ τόλμησαν να βαδίσουν σε μια ειρηνική διαδήλωση γιατί τόλμησαν ως, όπως οι γυναίκες να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο ή να προσπαθήσουν να ταξιδέψουν χωρίς ε, την έγκριση του συζύγου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα για τον 21ο αιώνα. Θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα σε οποιαδήποτε χώρα να τον κόσμο, αλλά δεν είναι αυτονόητα ούτε στη Σαουδική Αραβία μεταξύ άλλων χωρών. Είμαι πεπισμένη ότι το βραβείο Σαχάροφ για το Ραΐφ Μπαντάουι είναι ένα βραβείο ουσίας όταν μιλάμε για την ελευθερία σκέψης γιατί αν δεν είμαστε ελεύθεροι να σκεφτόμαστε και να εκφράζουμε τη σκέψη μας, πώς μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να δράσουμε σε μια κοινωνία, να την κάνουμε καλύτερη για την διαβίωση όλων και να δεχτούμε και τις διαφορές, τις διαφορετικές απόψεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε κοινωνία τα λόγια του συζύγου σας, οι πράξεις του, τα γραπτά του αποτελούν ένα σύμβολο ελευθερίας και δημοκρατίας. Όπου τον αποτολμά κανείς να μιλήσει, ακόμα και όταν ξέρουν ότι οι κυβερνώντες δεν, θα, ε, δεν αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, δείχνει το θάρρος. Το θάρρος του ανθρώπου πιστεύει στην αλλαγή του ε, κόσμου και θα ήθελα εν να σας συγχαρώ γιατί είχατε το θάρρος να ταξιδέψετε, να εξοριστείτε γιατί διαφορετικά θα διατρέχατε μεγάλο κίνδυνο με τα τρία σας παιδιά και σαν γυναίκα είχατε το θάρρος να τα κάνετε όλα αυτά. Το Σαββατοκύριακο είδαμε ότι για πρώτη φορά οι γυναίκες ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές και μερικές εξελέγησαν. όμως πώς στον 21ο αιώνα οι γυναίκες δεν μπορούν να εκλεγούν, δεν μπορούν να ψηφίσουν γιατί δεν μπορούν να βαδίζουν ελεύθερα που θέλουν χωρίς να έχουν το σύζυγο δίπλα ή οποιοδήποτε άντρα της οικογένειας. Γιατί θα πρέπει αυτό να είναι πρόβλημα σε οποιαδήποτε χώρα. Τη στιγμή που η νεωτερικότητα όπως τα αυτοκίνητα, τα κινητά, οι υπολογιστές υπάρχουν για να χρησιμοποιηθούν από τους πάντες. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο σύζυγός σας και εσείς ε, μιλήσατε για πρώτη φορά για τη σύγχρονη εποχή που δεν υπάρχει στη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης και λόγου. Και οι γυναίκες δεν μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Θα ήθελα να πω, όπως προελέχθη, η Σαουδική Αραβία είναι ένας μεγάλος γεωπολιτικός εταίρος. Θα θέλαμε να υπάρξει ειρήνη και εκεί, όπως και στη Συρία αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απλοί παρατηρητές των η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει αμάχους στην Ιεμένη και ελέγχει και εξάγει όπλα σε ένοπλες περιοχές. Έχει μεγάλη σημασία το ότι είσαστε εδώ αυτή την εβδομάδα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και πιστεύω ότι αυτό το βραβείο για το Ραΐφ Μπαντάουι δείχνει ότι θέλουμε να του αποδοθεί χάρη από το Ριάντ. Ελπίζουμε να ε, γίνει κάτι τέτοιο αυτές τις ημέρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καστάλντο. Φάμπιο Καστάλντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ειλικρινά και από τα βάση της καρδιάς μου καλωσορίζω την Ενσάφα Αϊντάρ που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι τιμή μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ΡΑΙΦ είναι σε απομόνωση αυτή τη στιγμή και έχει ξεκινήσει απεργία πίνες μετά από ε, φυλάκιση άδικη. Άδικη γιατί μετά από διάφορες παροδίες δικών ε, είπε αυτό που πραγματικά ήθελε. Ήψωσε μια φωνή ειλικρινή και δυνατή ε, και εξέφρασε το αναπαλατρίο το δικαίωμά του για να εκφράζει την άποψή του. Με μεγάλη πικρία ε, βλέπω τα βάσανα που τραβάει ο Ραΐφ. Δεν έπρεπε να είναι φυλακισμένο στο Ριάντ, θα έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας. Και υφίσταται μια ποινή που δεν είναι σωματική, είναι μια πραγματική θανατική ποινή σε δόσεις. Αισθάνομαι επίσης ε, θυμό γιατί και ο Ραΐφ και άλλοι που είναι φυλακισμένοι, ακριοτριάζονται, ε, φυλακίζονται, μαστιγώνονται, ακόμα και αν είναι ανήλικοι, ε, τα, λαμβάνουν, τα, τα, τα, υφίστανται αυτά σε μια χώρα η οποία είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βεβαίως είναι ένα καλό βήμα αυτό το βραβείο, αλλά δεν αρκεί. Είμαστε μία αγορά πολλών εκατομμυρίων καταναλωτών ε, και εμείς θέλουμε να αγοράζουμε και εκείνοι να ε, πολλούν. Ωστόσο, η ζωή μας είναι, η σχέση μας συγγνώμη, με τη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική από ότι με άλλες χώρες. Ε, ε εμείς εξάγουμε ε, όπλα. Ε, κάνουμε μεγάλες συμφωνίες με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ε, αγοράζοντας φθηνό πετρέλαιο. Και γνωρίζουμε ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πίσω από καταστροφές και θανάτους κατά χιλιάδες όπως στην περίπτωση της Ιεμένης. Ξέρουμε ότι διώκουν γυναίκες και παιδιά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ε, ότι διαρκώς ε, τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, των παιδιών ε, καταπατώνται. Όχι, δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε με ένα βραβείο Ζαχάροφ όλη αυτή την κατάσταση εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να συμφωνήσω με συμφωνίες εμπορικές με, οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε αντίτιμο. Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε αυτά που δεν είναι δυνατόν να ανεχτεί ένας άνθρωπος. Ο Ραΐφ δεν, και όχι μόνο αυτός θα πρέπει να ελευθερωθεί, να γυρίσει στη θαλπορή της οικογένειάς του και της γυναίκας του, αυτός και όλοι οι υπόλοιποι. στο όνομα μιας ε, λέξης που είναι η δικαιοσύνη που πολύ συχνά όλοι λησμονούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Χάινταρ. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ελευθερία και χωρίς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την ελευθερία έκφρασης. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τιμήσουμε για το θάρρος του και για την ελευθερία έκφρασης του τον Ραϊφ Παντάου αλλά και εσάς για το θάρρος σας λυπούμεθα πολύ που δεν μπορεί να έρθει σήμερα να πάρει αυτή την εβδομάδα ο ίδιος ε, στο Στρασβούργο το βραβείο του Ελπίζουμε όμως ότι θα απελευθερωθεί και θα μπορέσει παρόλα αυτά να έρθει. Και πραγματικά στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για να ενισχύσετε την ελευθερία έκφρασης. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σλίτς, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Κυρία Χάινταρ, ξέρω ότι με κυρία Λαμπρινή, σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα και εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά μπορούμε από κοινού σήμερα να δούμε το αποτέλεσμα κάποιων από τις ε, δράσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς γίνεται σήμερα σε κάποια δικτατορικά καθεστώτα. Ιδιαίτερα για μας ε, που γνωρίζουμε ότι σε πολλές χώρες όπως η Ανατολική Γερμανία αυτή η κατάσταση πριν από λίγο καιρό υπήρχε και ο σύζυγός σας σήμερα ζει μια κατάσταση την οποία γνώρισαν πολλοί στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν σήμερα να στηρίξω τις προσπαθειές σας, να χαιρετήσω το θάρρος σας και αυτό του συζύγου σας και να πω ότι δεν είναι η μόνη χώρα η Σαουδική Αραβία στην οποία παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι εξαιρετικά σκληρή η ποινή του και ξέρουμε ότι σήμερα βρίσκεται απομονωμένος και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Είναι λοιπόν ε, μια κατάσταση που εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να την παρατηρούμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να επιθύσουμε περισσότερο την προσοχή, τι ξέρετε εσείς, ξέρω ότι ο σύζυγός σας πραγματικά υποφέρει σωματικά, ψυχικά, σας ε, ευχόμαστε και ελπίζω να μπορέσετε να του περάσετε αυτό το μήνυμα κουράγιο, δύναμη και ελπίζω πολύ σύντομα να τον συναντήσετε, να απελευθερωθεί και να ξαναβρει τους δικούς του. Γιάννα Γκόμες. Πολύ σύντομα. Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε σήμερα εδώ από τον Ιανουάριο, όπως είπε και ο Ρίτσαρτ, Θελήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Λίγοι είναι συνάδελφοι που σας μίλησαν ήδη σε μια βίντεο συνδιάσκεψη που είχαμε οργανώσει. Και θεωρούμε ότι το βραβείο Ζαχάροφ αποτελεί μία από τις εκφράσεις υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την εκτίμησή μας σε σας προσωπικά και στις γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία. Όταν επισκέφτηκα τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγα χρόνια, συνάντησα γυναίκες όπως ε, αυτές τις 17 που για πρώτη φορά ήταν υποψήφιες για να εκλεγούν ε, στις δημοτικές εκλογές ε, της χώρας σας. Και βεβαίως ξέρουμε ότι αυτοί που πραγματικά φυλάνε τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία δεν είναι οι σύζυγοι τους, οι πατέρες τους και τα αδέρφια τους. Εσείς είστε οι πραγματικοί φύλακες. Εσείς φυλάτε την ελευθερία. Και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι παίζουν ένα ρόλο φύλακα για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας πραγματικά, ουσιαστικά περιορίζουν την ελευθερία τους και παραβιάζουν ε, τις θεμελιώδεις ε, ελευθερίες και αξίες, την αξιοπρέπεια των γυναικών. Σήμερα δεν μπορεί λοιπόν ο σύζυγός σας να έρθει εδώ για να πάρει το βραβείο του, αλλά αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές ε, στο παρελθόν άτομα ήταν στη φυλακή, βασανίστηκαν και τελικά μπόρεσαν και χάρη ίσως και στο βραβείο Ζαχάροφ να απελευθερωθούν. Υπάρχουν σήμερα σιήτες οι οποίοι συνεχίζουν να υποφέρουν, να καταδιώκονται, να είναι φυλακισμένοι και να εκτίουν πολύ αυστηρές ποινές. Ελπίζω λοιπόν η κατάσταση αυτή να αλλάξει. Εμείς σαν κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και για τον ε, Παλαιστίνιο ποιητή, τον Άσο Αφάγετ αλλά και άλλους, οι οποίοι και στην Σαουδική Αραβία και αλλού βρίσκονται στη φυλακή. 150 άτομα εκτελέστηκαν φέτος, όχι μόνο στη Σαουδική Αραβία, στο Γεμέν, στο Μπαχρέιν, κάτι που έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για όλη την περιοχή. Σήμερα βλέπουμε τους ε, τσιχάμπι, τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους Ισλαμιστές οι οποίοι τον απειλούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς, οι κυβερνήσεις μας, να έχουν εμπορικές συναλλαγές με αυτά τα καθεστώτα. Ο τελευταίος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Χάινταρ. Είμαστε πολύ ευτυχείς που είστε σήμερα εδώ. Εγώ ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, που πήγε στη Σαουδική Αραβία και μπόρεσα να συναντήσω εκπροσώπους ε, φορέων ε, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι μεγάλη η λύπη μας που σήμερα δεν έχει απελευθερωθεί ο Ραϊφ Μπαντάουι. Κάτι το οποίο θα ήθελα σήμερα να αναφέρω είναι το θέμα της παιδείας και δεύτερον το θέμα της δικαιοσύνης. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία έτσι ώστε να υπάρξει μία πιο συνεκτική πολιτική εντός και εκτός των συνόρων της Σαουδικής Αραβίας. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερος διάλογος. Είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος. Ήταν και στο παρελθόν και θα παραμείνει και στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Αραβίας. Ήταν πολύ σημαντικές και οι εκλογές που έλαβαν χώρα εχθές. Ελπίζω λοιπόν ο διάλογος μεταξύ της χώρας σας και, της Οδικής, ε, και της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αραβίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθεί και θα μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών, οι οποίες πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην πολιτική και στη δημόσια ζωή και ελπίζω να επιταχυνθεί η διαδικασία απελευθέρωσης των γυναικών στην Σαουδική Αραβία. Κάνω μια έκκληση γιατί πραγματικά θα πρέπει η κυβέρνησή σας, η βασιλική οικογένεια να δείξουν συμπόνια. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα του προφήτη Μοχάμετ Συμπόνια για όλη την ανθρωπότητα. Ελπίζω πολύ σύντομα να απελευθερωθεί λοιπόν ο Ραΐφ Παντάουι. Θα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χαϊντάρ, ακούσατε τους συναδέλφους από πολλές διαφορετικές πολιτικές ομάδες, χώρες. Βεβαίως και διαφωνούμε σε πολλά, αλλά όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες, είμαστε όλοι ενωμένοι. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να σας στηρίξουμε, να εκφράσω για άλλη μια φορά την υποστήριξή μας. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Τα λόγια σας ε, μου δίνουν ελπίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας. Ε, θα ήθελα να κάνω όμως δύο σχόλια. Ο Ραΐφ δεν βρίσκεται απομονωμένο σε ένα κελί έχει επανέλθει σε μία άλλη φυλακή την προηγούμενη Πέμπτη και πιστεύουμε ότι ο φάκελός του έχει πλέον αρχιοθετηθεί. Πρόκειται για μία φυλακή εκείνων όπου η περίπτωσή τους έχει τελεσιδικήσει. Βρίσκεται σε μία φυλακή εκεί κοντά στη Τζέντα, δεν είναι πλέον στο Ριάντ. Η απεργία πείνας άρχισε, την άρχισε την τρίτη την απεργία πείνας έτσι ώστε να επανέλθει στην φυλακή, να μεταφερθεί στη φυλακή όπου ήταν πριν και πριν από την απονομή του βραβείου είχα την ελπίδα να ε, απελευθερωθεί ο Ραΐφ μετά μου ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση ότι ασκούσε πίεση για την απελευθέρωση του Ραΐφ και ξαφνικά έμαθα ότι ο Ραΐφ μεταφέρθηκε σε μία άλλη φυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ για την απονομή του βραβείου. Έχει μεγάλη σημασία για μας. Πιστεύω να έχει αξία και έμπρακτα για την απονομή χάριτος στο ΡΑΙΦ και ότι θα έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες να ξαναειδωθούμε. Ελπίζω να είναι σε λίγες μέρες στο σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Elena, final word. Η Ελένα. Όχι, δεν έχω τίποτα να πω. Σας ευχαριστώ όλους και θα παρακολουθήσουμε την απονομή την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι που παρευρεθήκατε εδώ. Ε, υπάρχει ένα δείπνο για τους συντονιστές και τους προέδρους. Ευχαριστούμε κυρία Χαϊντάρ που ήρθατε εδώ απόψε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Σταύρο. Ε, έχεις μία μεγάλη εβδομάδα μπροστά σου γεμάτη δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.